με ενημέρωσε ότι δεν έχουν εγερθεί αντιρρήσεις στην σύσταση της απόφασης της Επιτροπής Απασχόλησης σχετικά με την απόφασή της να μην γύρει αντιρρήσεις σε σχέση με μια κατεξουσιοδότηση πράξη. Εάν εντός 24 ωρών μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 μέλη δεν εγείρουν οποιαδήποτε αντίρρηση, αυτή η σύσταση θα θεωρηθεί εγκεκριμένη, διαφορετικά θα ε, υπάρξει ψηφοφορία. Είναι στη διάθεσή σας ε, η ε, πρόταση αυτή στο, στην ιστοσελίδα. Επίσης, η